το άρθρο 78 του κανονισμού μας σε ε, κοινή πράξη με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου θα υπογράψουμε τις πράξεις νομοθετικής διαδικασίας, κοινής νομοθετικής διαδικασίας ε, που προβλέπονται